ήδη τώρα έχουν κερδίσει τμήματα της αγοράς εις βάρος ε, των ευρωπαϊκών εταιριών παρά των διαρθρωτικών αλλαγών και της αύξησης παραγωγικότητας που έχουν επιτύχει οι δικές μας εταιρείες. Εφόσον λοιπόν υπάρχει τέτοια στρέβλωση του ανταγωνισμού, τότε πρέπει εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> να δράσουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένα μέτρα, κατά τον, ε, του dumping των επιδοτουμένων εταιριών, αλλά και με τις κατάλληλες ενέργειες όταν ε, οι εταιρείε μα σε άλλα μέρη του κόσμου για τα δικαιώματα προσγείωση για τι υπηρεσίε εδάφου υφίστανται διακρίσει. Ο κανονισμό 868 επιτρέπει ήδη να ξεκινούν έρευνε για τα θέματα αυτά. Όταν ε, υπάρχει κίνδυνο ζημία ή αναγγέλλονται διακρίσει, πριν δηλαδή προκύψουν ακόμη όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γεγονό ότι μπορεί να δράσει ακόμη και όταν υπάρχει απειλή έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Γενική Διεύθυνση Τραν μπορεί να δράσει όταν υπάρχει μόνο και κίνδυνος. Αυτό οφείλεται στην ενέργεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που το επιβάλαμε κατά τους τριμερείς διαλόγους. Και μόνο έτσι Αποκτά δόντια ο κανονισμός 868. Είναι πραγματικός αποτρεπτικός μηχανισμός. Αν πάει καλά, ίσως να μην χρειαστεί να τον εφαρμόσουμε ποτέ. Ο κανονισμός αυτός είναι και ένα διπλωματικό μέσο λοιπόν για την Ευρώπη και για τα κράτη-μέλη που από μόνα τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις διακρίσεις. Εάν όμως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση όλων των κρατών μελών επιχειρεί να αντιδράσει, τότε έχουμε παγκόσμια επίδραση και στον τομέα των ε, αεροπορικών μεταφορών. Η απάντησή μας στο σύνθημα America First, Gulf Airlines First, China First είναι Europe Together. Η Ευρώπη από εκείνο ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το καλό κείμενο που προτείνει. Ευχαριστώ το Συμβούλιο για τι δύσκολε αλλά τίμιε διαπραγματεύσει και ευχαριστώ εσά, συνάδελφοι, που εδώ βοηθήσατε αποφασιστικά. Έχουμε τώρα ένα καλό βασικό κείμενο για μια Ευρώπη που να μπορεί να περασπίζει τα συμφέροντά τη άλλο ένα ε, στοιχείο στην οικοδόμηση μιας ισχυρής Ευρώπης που αντιστέκεται. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Και τώρα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπο Έτιγκερ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Εκπροσωπώ τον συνάδελφο Μπούλτ, ο οποίο δυστυχώ είναι ασθενή. Αλλά ευχαριστεί πολύ που σήμερα Ε, γίνεται αυτή η συζήτηση εδώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Πίπα. που υπέβαλε την έκθεση αυτή στο Κοινοβούλιο και ευχαριστώ και την αρμόδια επιτροπή που επέφερε ε, σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενο και η οποία έκανε ουσιαστική δουλειά λοιπόν. Ευχαριστώ και τους Κιώδης που και αυτοί συνέβαλαν ιδιαίτερα. Η έγκριση του νέου κανονισμού για την διασφάλιση ισοτήμου ανταγωνισμού στις ε, αεροπορικές μεταφορές είναι μεγάλο στοιχείο τη ε, στρατηγική μα για τι αεροπορικές μεταφορέ. Ξεκινήσαμε πριν από τέσσερα χρόνια αυτή την προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα έχουμε πλέον, πλέον μάλλον, την νομική βάση γι' αυτό. Αυτό ο κανονισμό είναι βασικό στοιχείο των μέσων που διαθέτουμε για ισότιμο ανταγωνισμό στις ευρωπαϊκές ε, αεροπορικέ μεταφορές και στην εξωτερική μας πολιτική έναντι άλλων χωρών όπου θέλουμε να υπάρχει ισότιμο ανταγωνισμός. Οι αλλαγές στον κλάδο αυτών για τη μεταφορά και των ε, επιβατών και προϊόντων είναι ουσιώδης. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και τα κατάλληλα μέσα που να μπορούν να λειτουργούν ούτως ώστε όλες οι αεροπορικές εταιρείε και επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον κλάδο να μπορούν να εργάζονται σε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού. Να είναι εγγυημένο αυτός ο ισότιμο ανταγωνισμό. Αφορά τις πτήσεις ε, και προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός αυτός. Και εδώ έχουμε και τις εταιρείε μας που εδρεύουν στην Ένωση και ανταγωνιστές που ε, έχουν την έδρα τους εκτός τον ε, αποδεχόμεθα και τον εκτιμούμε αυτόν τον ανταγωνισμό. Και το θέμα είναι και πώς θα γίνονται σωστά και αεροπορικέ συνδέσεις. Ποιος θα τις εγγυάται. Για τις πτήσεις προς την Ένωση, οι αεροπορικές εταιρείε των τρίτων χωρών έχουν τη δική μας εγγύηση. Ότι υπάρχουν ε, ευρωπαϊκοί κανόνες που ισχύουν και για αυτούς. Όπως ακριβώς για τις ε, δικές μας εταιρείε. Εμείς, σαν Ένωση, θέλουμε όντως ισότιμο ανταγωνισμό με ταυτόσιμες συνθήκε. Και τον εγγυόμεθα, αλλά διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς δεν αλλάζει, αλλά αντίθετα και ενισχύεται η διακριτική μεταχείριση που υφίστανται οι εταιρείε μας έναντι των εταιρεών εκτός Ένωσης. Και αντιμετωπίζουν ε, διακρίσεις λοιπόν και βρίσκονται σε μειονεκτούσα θέση. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη δική σας στήριξη θεωρούμε ότι ο ανταγωνισμός πρέπει να υπάρχει σε ένα πολυμερές πλαίσιο και με παγκόσμια εναρμονισμένες συνθήκες. Αλλά ούτε ο ΠΟΕ, ούτε οι οδηγίες του ΙΚΑΟ, ο Διεθνής Οργανισμός της ε, Πολιτικής Αεροπορίας, δεν είναι ρεαλιστικές ούτε τώρα ούτε για το μέλλον. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να δράσουμε. Αποφασίσαμε και θέλουμε να έχουμε ε, συμφωνίε με τρίτε χώρε που να διασφαλίζουν αυτόν τον αγωνισμό. Μέχρι τώρα οι μεταξύ Ένωση και τρίτων χωρών βασίζονται σε μεμονωμένε συμφωνίε, δηλαδή συμφωνίε μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών με τι τρίτε χώρε. Αλλά αν βρούμε ω 28 ή 27 έναν των τρίτων, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και γι' αυτό με τον κανονισμό που συζητάμε τώρα, η Ένωση δημιουργεί τη βάση για αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Για να δράσουμε προ το συμφέρον των κρατών μελών, των πολιτών μα, για να υπάρχουν θέσει εργασία, για να εξακολουθούν να λειτουργούν οι εταιρείε αυτέ. Ούτω ώστε οι αθέμητε πρακτικέ να σταματήσουν και με το μέσο αυτό να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε τέτοιε αθέμητε πρακτικέ. Ο κανονισμό αυτό που έχετε ενώπιον σα σήμερα και στη διαμόρφωση του οποίου παίξατε θεμελιώδη ρόλο είναι πολύ πιο βασικός από τον προηγούμενο που ήταν από το 2004 και ο οποίος ε, στην πραγματικότητα δεν μπορούσε να εφαρμοστεί και αποδείχθηκε αναποτελεσματικός. Ο κανονισμός που προτείνουμε τώρα ασχολείται με τις ιδιαιτερότητες ε, του ε, τομέα αυτού σήμερα και θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό οι συμφωνίες αυτές να εξακολουθούν να συμφωνούνται με τις τρίτες χώρες. Επιδιώκουμε πάντα το διάλογο και συμβαστικές λύσεις. Τα προτιμούμε αυτά έναντι μονομερών λύσεων. Οπότε θεωρώ ότι σήμερα είναι σημαντική μέρα για τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ της, ε, του αεροπορικού κλάδου στην Ένωση και των ε, εταιριών εκτός Ένωσης και των πολιτών μας που θέλουν να πάρουν το αεροπλάνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, τώρα για την ε, ΕΚΟΝ, ο κύριος Τρεμόσα, παρακαλώ. Καλώ ήρθατε κύριε Πίτρο πάλι μια φορά εδώ. Αυτή συνάδελφοι, σε ένα πλαίσιο υψημένου ανταγωνισμού μεταξύ των αερομεταφορέων σε παγκόσμιο επίπεδο, ο δίκαιο ανταγωνισμό, ο θεμητό ανταγωνισμό και οι ίδιοι κανόνε είναι σημαντική αρχή την οποία θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει. Το να ζητούμε ε, να ισχύουν οι ίδιοι κανόνε ε, για όλου του ε, αερομεταφορεί δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται προστατευτισμό. Ε, όπως ε, ζητούμε από πολλούς αερονοφερείς να αναδιαρθρωθούν και να σταματήσουν να εξαρτώνται από εξωτερική χρηματοδότηση και από επιδοτήσεις, έτσι ζητούμε, ζητώ αυτή τη στιγμή και ε, να ισχύσουν ήδη οι κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει 550 εκατομμύρια ενδεχόμενων επιβατών ξένες εταιρείε από την Ασία για παράδειγμα χρησιμοποιούν την Ευρώπη ως ε, ε, hub και να γεμίσουν τα αεροπλάνα τους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε τη ρήτρα της ε, οικονομικής διαφάνειας με τις επενδύσεις τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκές αερομεταφορές αν λαμβάνουν επιδοτήσεις, γιατί θα πρέπει να ε, τους δίνεται τη δυνατότητα να ελέγχουν ευρωπαϊκές ε, εταιρείε αερομεταφορών. Δεν είναι θεμητός ανταγωνισμός αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τις παρεμβάσεις εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Ξεκινάμε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και δίνω το λόγο στον κύριο Βάντεν Κάμπα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Καλωσορίσατε στην Ολομέλεια. Ελπίζω ότι θα διαβιβάσετε τις ευχές μας στην Βιολέτα Μπούλτσο. Από ό,τι φαίνεται βελτιώθηκε η υγεία της, αυτό έμαθα σήμερα. Σε κάθε περίπτωση διαβιβάστε τις τις ευχές μας. Να ευχαριστήσω επίσης τον εισηγητή, τον συνάδελφο Μάρκους Πίπερ, για την εξαιρετική του εργασία και τη σκληρή δουλειά που έκανε προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκθεση αυτή. Το ζήτημα αυτό ολοκληρώθηκε υπό την Αυστριακή τότε Προεδρία και είναι περίεργο ότι εμείς συζητάμε τώρα μόνο αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου. Κύριε Πρόεδρε και ο Πρόεδρος Επιτροπής ΕΚΟΝ αλλά και ο Επίτροπος το είπανε, πρόκειται για να ζήτημα, μια πρωτοβουλία που είναι πάρα πολύ σημαντική και σε διεθνές επίπεδο. Και τους τελευταίους μήνες έχει γίνει ακόμα πιο σημαντική η πρωτοβουλία αυτή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες συναδιόμενες εθνικιστικές στάσεις παντού στον κόσμο και εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι οι διεθνείς αεροπορικές μεταφορές θα παραμείνουν ανοιχτές. Πιο εύκολο να το λέει κανείς αυτό θεωρητικά από ότι να το διασφαλίζει στην πράξη. Το να καταφέρουμε όμως να κρατήσουμε ανοιχτή την διεθνή αεροναυτιλία στα πλαίσια μιας θεμητής δίκαιης αγοράς, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς υπάρχει με ένα μεγάλο ποσοστό αθέμητο ανταγωνισμό αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν ακόμα και παράνομε κρατικέ ενισχύσει. Και ξέρετε, δεν μιλάμε εδώ πέρα μόνο για τα κάψιμα όπω η κεροζίνη ή για τι αραβικέ χώρε Έχουμε και την Κίνα, το Χονγκ Κόνγκ, ακόμα και τη Σιγκαπούρη που εμπλέκονται σε τέτοιες αθέμητες πρακτικές και αντιμετωπίζουν σε όλες τις αγορές αυτές αθέμητο ανταγωνισμό οι δικές μας ευρωπαϊκές εταιρείες. Ελπίζω ότι μέσω της έκθεσης αυτής θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την κατάστασή τους και να διασφαλίσουμε για τις εταιρείες αυτές συνθήκες πιο θεμητού ανταγωνισμού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματος τώρα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών το λόγο έχει ο κύριος Πρόης. Παρακαλώ. Η κυρία Πρόης, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι βάση τη ευημερία μα στην Ένωση είναι ο ισότιμο ανταγωνισμό και η κοινωνική ισότητα. Αυτό ισχύει και για ε, τι διεθνεί αεροπορικέ μεταφορέ. Ω νομοθέτε, πρέπει να προσφέρουμε στι ε, εταιρείε και στου εργαζόμενου προστασία από αυτέ τι αθέμητε πρακτικέ, για να έχουν υψηλού επίπεδου θέσει εργασία στην Ένωση. Γιατί ζούμε σε μια εποχή εμπορικών πολέμων. Μόνο με αρκετά αποτρεπτικά όργανα μπορούμε να επιζήσουμε στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και να επιβάλλουμε δίκαιου κανόνε για την Ευρώπη. Γι' αυτό χρειαζόταν αναθεώρηση του κανονισμού 868. Ήταν απόλυτα αναγκαία και επίγουσα. Όμω από πλευρά του Συμβουλίου δεν βλέπουμε να είναι σωστά τα πράγματα. Είναι πολύ περίεργα αυτά που βλέπουμε. Υπάρχει μια ομάδα κρατών μελών που είναι κατά αυτή τη πρωτοβουλία, κατά του να έχουμε αυτό το προστατευτικό μέτρο. Δεν θέλουν να υπάρχουν αυτά τα μέτρα και μάλιστα δίνουν και παράνομε κρατικές επιδοτήσεις. Μόνο για λόγους ε, ιδεολογικής ε, πίστης στον ε, κανόνα των ελευθέρων αγορών. Για μας το βασικό είναι να είναι ρωμαλαίο το κείμενο αυτό, να προστατεύει τι εταιρείε μας. Έχουμε, θα έχουμε έτσι ένα αποτελεσματικό μέσο κατά των επιζημίων επιδοτήσεων από πλευρά τρίτων χωρών. Δεν πρόκειται για προστατευτισμό, εις βάρος των επιβατών ε, ή ε, εις βάρος της δυνατότητας συνδέσεων, δηλαδή διαδρομών. Κανένας δεν πρέπει να φοβάται τον ελεύθερο ανταγωνισμό, αλλά οι ομάδες νομίζω ότι επέτυχαν ένα σωστό και ε, ευρέως στηριζόμενο συμβασμό και ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Πίπα και τους συνεργάτες του, αλλά και τους άλλους που έπαιξαν ρόλο. Ευχαριστώ για την επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρο Και τώρα για τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστές η κυρία Φώστερ, 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, έχουν περάσει πολλοί χρόνος από τότε που πρώτο ανταλλάξαμε απόψη αυτό το θέμα. Το αρχικό κείμενο της ε, Κομισιόν ε, έλαβε μια προσέγγιση προστατευτική που θα επέτρεπε στην Κομισιόν να επιβάλλει ποινές σε αερομεταφορείς τρίτων χωρών πριν να γίνει ολοκληρωμένη εξέταση των παραπώνων. Αυτό θα ήταν πραγματικά πολύ αρνητικό σημάδι για τους εταίρους μας και θα μας ζημιώνε παγκοσμίω και σε ό,τι αφορά τη φήμα μας και σε ό,τι αφορά τη συνδεσιμότητά μας. Επίσης το κείμενο επέτρεπε ε, μία ανταγωνιστική αερομεταφορή στην Ευρώπη να ε, κάνουν αγωγές εναντίον ε, ανταγωνιστών τους. Προφανώς είναι σωστό να αντιμετωπίσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά όχι ζημιώνοντας τη δυνατότητα των επιβατών να επιλέξουν και αυξάνοντας το, τα κόστη και τον, την τιμή των εισιτηρίων. Μετά τον τριμερή διάλογο όμως μπορώ να στηρίξω την τελική συμφωνία Καταρχήν διότι διευκρινίζει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, όπως για παράδειγμα τη ρύθμιση των διαφορών μέσω διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες, ε, αλλά και για άλλους λόγους. Ε, πιστεύω ότι το κείμενο είναι ισορροπημένο και θα επιτρέψει ε, να αυξηθεί η αγορά και να γίνουν πιο ισχυρές οι σχέσεις με τρίτες χώρες. Αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, να πω ότι είναι η τελευταία μου μάλλον ομιλία στην Ολομέλεια. Η πρώτη μου ήταν το 1999 και να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους ε, διερμηνείς και εδώ και στις Βρυξέλλες, τη Γραμματεία και όλο το προσωπικό του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στήριξή τους και τον επαγγελματισμό τους. Σε εύχομαι καλή επιτυχία στο μέλλον σε ό,τι επιχειρήσουν. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφε. Εξ ονόματος τώρα της ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, ο Αντιπρόεδρος Τελίτσκα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Τζάκη, που ήταν εξαιρετική συνάδελφος και πραγματικά ήταν πάντα ευχαρίστη για μένα να συνεργάζομαι μαζί σου. Σε εύχομαι ότι καλύτερο. Όσον αφορά τώρα αυτή την πρόταση κανονισμού, τρία πράγματα θα ήθελα να πω. Πρώτον, αποτελεσματικότητα, συμπληρωματικότητα και τρίτον, διάλογος, αποτελεσματικότητα. Γιατί επιτέλους έχουμε ένα μέσο το οποίο έχει έναν εμπορικό αμυντικό χαρακτήρα, αλλά δηλαδή δίνει επίση και τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξάγει έρευνε αν υπάρχουν εύλογοι λόγοι βάσει καταγγελιών και θα μπορεί βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από μόνη τη με δική τη πρωτοβουλία να κάνει έρευνε. Αποτελεσματικότητα, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρειάζεται πλέον να περιμένει από έναν ευρωπαϊκό αερομεταφορέα να επηρεαστεί, να ζημιωθεί, αλλά μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προληπτικά να λάβει δράση αν φανεί τελικά ότι υπάρχει κάποια ένδειξη ή ακόμα και απειλή επιζήμιας αθέμητης συμπεριφοράς. Και έπειτα έχουμε και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάγραμμα και για τις έρευνες και για τον τερματισμό των ερευνών. Και έχουμε επίσης και τη δυνατότητα να συντομεύσουμε το χρονικό αυτό πλαίσιο αν ισχύουν συνθήκες της έκτατης ανάγκης και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, γιατί αυτή τη στιγμή μέσω της νέας αυτής πρόθεσης κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα κατά αερομεταφορέων. Τώρα, συμπληρωματικότητα. Θεωρώ ότι σε συνεργασία με τις υπόλοιπες διμερείς συμφωνίες που έχουμε συνάψει, που θα συνάψουμε, έχουμε ένα πολύ πιο σφαιρικό ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο θα μας επιτρέψει να συμπληρώσουμε τις διμερείς μόνο τώρα προσπάθειες για να επιλύσουμε τις διαφορές. Τώρα διάλογος. Διάλογος και διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη θα προβλέπετε πάντα προς το συμφέρον το ευρωπαϊκό. Θα έχουμε διάλογο επίσης με τους συμμετέχοντες. Αυτό προβλέπεται από τους μηχανισμούς διαλόγου. Και τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται δεόντως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Δεν μιλάμε λοιπόν για προστατευτισμό, αλλά μιλάμε για ένα πολύ καλό εργαλείο που θα έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματος των Πρασίνων τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντέλη. Έχετε το λόγο, Καριμά. Θα ψηφίσουμε ένα από τους τελευταίους ε, κανονισμούς ε, κατά ε, τη διάρκεια της θητείας μας για τον τομέα των αερομεταφορών. Ο θέμητος ανταγωνισμός είναι πραγματική μάστιγα σε αυτόν τον κλάδο. Για παράδειγμα, οι, χώρες του, οι εταιρείε του κόλπου που χρηματοδοτούνται και επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις τους για να πληρώσουν τα τέλη αεροδρομίου και την κυροζήνη τους. Ε, ε, χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν καταστρέφει με αυτόν τον τρόπο γιατί οι δικές μας εταιρείε δεν μπορούν να ακολουθήσουν και γι' αυτό το λόγο πολλοί εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους. Αυτή η μάστιγα δημιουργεί και άλλη μια μαστιγά. Ενώπιον αυτού του αθέμητου ανταγωνισμού ε, δημιουργεί μια καινούρια, δημιουργεί καινούριε διαδρομέ περισσότερων χιλιόμετρων για να ενωθεί η Ευρώπη με την Ασία μέσω των χωρών του κόλπου. Και αυτό δημιουργεί αύξηση και τη μόλυνση. Συνεπώ, έχουμε και κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που είναι αλληλένδετα. Ως ε, πολίτες, καταναλωτές και εργαζόμενοι είμαστε όλοι θύματα αυτής της κατάστασης. Σας θυμίζω ότι ο κλάδος αυτός αντιπροσωπεύει το 3% των, παγκόσμιων εκπομπών. Ε, είναι σαν να λέμε εκπομπές όλης της Γερμανίας. Και τι κάνει αυτό το κείμενο για να αντιθώ στην κατάσταση. Πολύ λίγα πιστεύω, φοβάμαι. Γιατί το πρόβλημα είναι βαθύ ε, είναι τεράστια η πρόκληση της αναδιάρθρωση του κλάδου. Το είδαμε στις ε, συμφωνίε του Παρισιού του 2015. Ο κλάδος αυτός είχε εξαιρεθεί πλήρω των διαπραγματεύσεων. Αυτό όμω που πραγματικά με λυπεί είναι ότι βλέπω πως σήμερα η Ευρώπη υφίσταται ένα, ένα παγκόσμιο σύστημα το οποίο δεν αναλαμβάνει τι ευθύνε του για την ε, κλιματική, ε, αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε προτείνει ε, το φόρτς και άλλες ε, λύσεις ε, τις οποίες αρνούνται. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε ο κλάδος να αυτοαναδιαρθρωθεί, να αυτομεταρρυθμιστεί. Εμείς οι ονομοθέτης θα πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ο τομέας των αερομεταφορών είναι μια πρόκληση, το είπαμε, είναι μια οικονομική πρόκληση, είναι μια κοινωνική πρόκληση, αλλά κυρίως είναι μια κλιματική πρόκληση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σιγεί μπροστά σε αυτή την πρόκληση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο τώρα εξ ονόματος της ομάδας Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, έχει ε, ο κύριος Πιμέντα Λόπες. Ζωάο, έχει το λόγο. Αυτή η πρόταση κανονισμού δημιουργεί διάφορα θέματα που μας ε, ανησυχούν. Ε, στο πλαίσιο της ενίας αγοράς, στο πλαίσιο της διατηρικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί τη συγκέντρωση σε ένα κλάδο, δημιουργεί μονοπόλια σε αερομεταφορές και είναι μια στρατηγική η οποία θα οδηγήσει σε καταστροφή ε, εταιριών που τροφοδότησαν την όλη διαδικασία ιδιωτικοποίηση ε, σε ευρεία κλίμακα. Είναι μια διαδικασία η οποία δημιουργεί σημαντικές ζημίες για τις χώρες αλλά και για τους εργαζόμενους που βλέπουν τα δικαιώματά τους, εργατισιακά τους δικαιώματα πλήττονται. Αυτός ο περίφημος περιβόητος ανταγωνισμός είναι στο κέντρο αυτής της πρότασης ε, που δημιουργεί μια διάκριση ανάμεσα στις, ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκές εταιρείες και στις μη ευρωπαϊκές εταιρείες που ανταγωνίζονται για την ίδια αγορά. Θέλουμε να ε, τεθούν προϋποθέσεις στην αδειοδότηση εταιριών οι οποίες λαμβάνουν ε, χρηματοδότηση και επιδοτήσεις από το κράτος. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Ε, με τον ίδιο τρόπο πανεμβαίνουμε και σε εθνικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργείται, συνεπώς, μια, δημιουργούνται λοιπόν εταιρείε ε, χαμηλού κόστους ε, που, ε, με χαμηλότερη ποιότητα και λιγότερα δικαιώματα στους εργαζόμενου. Αυτοί είναι λόγοι για να απορρίψουν αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματο της Ομάδας Ευρώπη Ελευθερίας και άμεση δημοκρατία το λόγο έχει η κυρία Αιούτο. Για ένα λεπτό, Ντανιέλ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπω το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τον θεμητό ανταγωνισμό, προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρήσεις χωρίς διακριτική μεταχείριση. Όμως, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αμοιβαιότητα από άλλες τρίτες χώρες και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις δικές μας τι να θεσπίσουν μέτρα για να ταχθούν κατά των αθέμητων πρακτικών. Υπάρχουν βέβαια κάποιες διμερείς συμφωνίες προσπαθούν να θεσπίσουν αυτά τα επαναρθωτικά μέτρα δεν λειτουργήσε αποτελεσματικά ο κανονισμό 868 και γι' αυτό το λόγο θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα κανονισμό πιο αποτελεσματικό όσον αφορά τι έρευνε, όσον αφορά τα επαναρθωτικά μέτρα, διότι α μην ξεχνάμε ότι ο ισχύων κανονισμό 868 ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε. Αν πραγματικά θέλουμε να προστατεύσουμε τη συνδεσιμότητα για του πολίτε μα και πραγματικά θέλουμε να έχουμε θεμητό ανταγωνισμό για του αερομεταφορεί μα, για τον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τα απαραίτητα μέσα ελέγχου. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο κύριος Σότσνιερ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κανονισμός αυτός της μας λέει ότι ο αθέμητος ανταγωνισμός βασίζεται σε κάποια πλεονεκτήματα, σε κάποιες επιδοτήσεις και ενισχύσεις που δίνουν οι κυβερνήσεις. Συμφωνώ με αυτό. Αυτό είναι όντως αθέμητος ανταγωνισμός. Αν παίρνετε χρήματα από τους φορολογουμένους και τα δίνετε σε έναν νερομεταφορέα γιατί τα χρήματα αυτά ουσιαστικά είναι ενέδο κλοπή στην περίσταση αυτή. Αλλά εμεί εδώ βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι κάνουμε. Εμεί επιδοτούμε τα πράγματα εδώ πέρα, μεταφορέ, γεωργία, του ίδιου φοιτητέ, μη κυβερνητικέ οργανώσει. Και νομίζω ότι επιδοτούμε και τις αεροπορικές μεταφορές. Πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε έδωσε την άδεια μάλλον στην Πολωνία να πάρει χρήματα από τους φορολογούμενους και να τα δώσει στον Εθνικό Αερομεταφορέα. Ανάλογα παραδείγματα έχουμε δει και σε άλλες χώρες, επομένως δεν νομίζω ότι μπορούμε να ερχόμαστε εμείς εδώ πέρα και να λέμε ότι δεν λειτουργούν καλά τα πράγματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι κατηγορούμε κάποιες εταιρείες ενώ κρύβουμε τις ίδιες τις δικές μας πρακτικές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Λούτς έχει τώρα το λόγο για δύο λεπτά. Η... Ευχαριστώ πολύ. Οι αερομεταφορέ ε, είναι βασικό τομέα για την ανάπτυξη τη ευρωπαϊκή οικονομία και υπάρχει τεράστια ανάπτυξη στον αριθμό πτήσεων και εντό ε, και από την Ένωση προ ε, άλλα μέρη. Είναι μια, μια αγορά που αναπτύσσεται με εκθετικό ρυθμό παρά τις πιέσεις που υπάρχουν ε, σε αυτήν την οικονομική δραστηριότητα που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση και τον ανταγωνισμό από χώρες της Ασίας. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείε αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό των εταιρεών του, της Μέσης Ανατολής που έχουν ε, τεράστιο κεφάλαιο στη διάθεσή τους και ε, δίνουν καταπληκτικές τιμές και πολύ πλούσια δρομολόγια και αποφεύ, δεν χρειάζεται να εφαρμόζουν τις ε, νομοθεσίες μας. Και αυτό σημαίνει ότι και αυτοί αναπτύσσονται δυναμικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη είναι αθέμητο ο ανταγωνισμό. Συμφωνώ με όλου του προηγούμενου ομιλητέ που είπαν που, ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλήγουμε σε, σε συμφωνίες με τις αναδυόμενες και στρατηγικές αγορές και όλα αυτά πρέπει να έχουν και μία ρήτρα δικαίου ανταγωνισμού. Χρειαζόμαστε ένα σωστό σύστημα αποζημιώσεων ούτω ώστε να υπάρχουν συνθήκε ισότιμου ανταγωνισμού για τι ε, αεροπορικέ μα εταιρείε. Και νομίζω ότι αυτό ο κανονισμό είναι ένα μέσο που θα ενισχύσει το βάρο μα σε αυτή τη διαπραγμάτευση και θα ενισχύσει και την ε, οικονομική αυτή δραστηριότητα. Ωστόσο, οι καταναλωτέ, οι επιβάτε ε, επιλέγουν κυρίω με βάση την τιμή του εισιτηρίου αλλά και με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών του παρέχονται πώς ε, θα περάσουν στην πτήση αλλά και το που πάνε, Ποιο είναι ο προορισμό. Εάν λοιπόν θέλουμε να στηρίξουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείε, τότε ε, θα βάλουν σε πρώτη γραμμή τον ε, επιβάτη. Και αυτό είναι κάτι που κανένας κανονισμός δεν μπορεί να στο επιβάλλει. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον κύριο Σόρνια. Την αδέχεστε, τη δέχεστε. Ε, λυπάμαι συνάδελφο Σόσνιερ, η συνάδελφο δεν δέχεται την μπλε κάρτα. Και τώρα τα παρντέλ. 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Πίπα, που κατάφερε να υπάρξει διοργανική συμφωνία για ένα τόσο σημαντικό θέμα για το μέλλον των ε, αερομεταφορών. Οι εταιρείε μας εντάσσονται σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο που ε, διασφαλίζει την σύνδεση της Ευρώπης με τον υπόλοιπο κόσμο και τις εσωτερικές συνδέσεις βέβαια. Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε τον πλάδο αυτό μέσω των αναγκαίων μηχανισμών και εργαλείων για να τιμωρούνται οι αθέμητες πρακτικές τρίτων χωρών. Παράλληλα βέβαια πρέπει να διασφαλίζονται επαρκείς συνδέσεις για τους επιβάτες, επαρκή δρομολόγια. Υπάρχουν βέβαια κάποιες κρατικές ενισχύσεις που μπορούν να στρεβλώσουν ιδιαίτερα τον ανταγωνισμό. Οι εσωτερικές τώρα πτήσεις πρέπει να διεξάγονται με βάση σωστές ηθίκες θεμητού ανταγωνισμού. Όμως αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχουν σωστέ συνθήκε εργασία για του εργαζόμενου στον τομέα αυτό, να προσφέρονται σωστέ υπηρεσίε στου επιβάτε και επίση να σεβόμαστε το περιβάλλον. Ω υπεύθυνοι για τα θέματα του τουρισμού, θέλω να στείλω μήνυμα στι ευρωπαϊκέ εταιρείε να προσέξουν τι δικέ του πρακτικέ, γιατί ορισμένε φορέ ε, οι ειδικέ του πρακτικέ ε, τι κάνει να χάνουν ε, τμήματα τη αγορά έναντι εταιρεών τρίτων χωρών. Αυτό που συστήνω λοιπόν είναι να προσέχουν γιατί πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επίπεδου αν θέλουν να προσελκύουν επιβάτες και η σχέση τιμής και ποιότητας υπηρεσιών πρέπει να είναι καλή. Η Ευρώπη πρέπει να είναι στην πρωτοπορία των παγκοσμίων αερομεταφορών όσον αφορά όλες τις προδιαγραφές ποιότητας. Βεβαίως και όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατών και τους όρους εργασίας στις εταιρείες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Παπαρντέλ, και τώρα ο κύριος ε, Λωτόφσκι. Ο ανταγωνισμός στις αερομεταφορές ε, είναι απαραίτητος και τον αναμένουν και οι καταναλωτές. Αλλά θα πρέπει να βασίζεται σε υγιείς αρχές που θα αποκλείουν τον αθέμητο ανταγωνισμό εκ μέρους τρίτων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτει εργαλεία αυτοπροστασίας έναντι του αθέμητου ανταγωνισμού από εταιρείε οι οποίες λαμβάνουν επιδοτήσεις, κρατικές επιδοτήσεις που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο κανονισμό είναι μια ευκαιρία να εκριζώσουμε τέτοιε ε, πρακτικές, οι οποίες τελικά ζημιώνουν τους ίδιους επιβάτες. Πάνω απ' όλα όμως, χρειαζόμαστε διεθνεί λύσει που θα αποκλείουν την χρήση ε, πρακτικών αθέμητου ανταγωνισμού στον κλάδο αυτό. Χρειάζεται να πιέσουμε περισσότερο Τρίτε χώρε με τι οποίε διαπραγματευόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς, αγαπητέ συνάδελφε. Περνάμε τώρα στη δικασία Catch the Eye. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο εδώ. Ξεκινάμε με τον κύριο Μαριά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο κανονισμός 868 είναι βέβαιο ότι πρέπει να εφαρμοστεί διότι μόνο έτσι θα σταματήσει ο αθέμητος ανταγωνισμός που γίνεται από εταιρείες τρίτων χωρών εταιρείες οι οποίες πραγματικά έχουν βρει την ευκαιρία λόγω και της απραξίας που υπήρχε στην ευρωπαϊκή ένωση να ανταγωνίζονται αθέμητα τις ευρωπαϊκές εταιρείες. όμως θα πρέπει και στο εσωτερικό στις εσωτερικές πτήσεις να υπάρχει ο ανταγωνισμός και ήθελα κύριε επίτροπε κύριε Έτιγκεν, να επισημάνω για άλλη μια φορά το θέμα με την εταιρεία την αεροπορική aegean η οποία είναι κυριολεκτικά μονοπόλιο στην ελλάδα και υπάρχουν πανάκριβα εισιτήρια από την κρήτη για να ταξιδέψεις αεροπορικά στην αθήνα πληρώνεις περισσότερα από ό,τι πληρώνεις το εισιτήριο από την αθήνα για το βερολίνο. αυτό ισχύει επίσης με τα ακριβά εισιτήρια και για τα νησιά του αιγαίου. πρέπει να υπάρξουν μέτρα και στα θέματα αυτά το έχω καταγγείλει από τον νοέμβριο του 2018. δεν έχω πάρει απάντηση. δεν μπορεί να έχουμε αυτό το καθεστώς μονοπωλίου στην ελλάδα με πανάκριβα εισιτήρια από την κρήτη προς την ηπειρωτική ελλάδα από τα νησιά προς την ηπειρωτική ελλάδα. ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σέτεριτς τώρα για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ανησύχησα όταν ο εισηγητής έρθα μας λέει ότι από κοινού θα καταφέρουμε να τα βάλουμε με την Κίνα κτλ. Και άρχισε να μιλάει έπειτα βέβαια για την διασφάλιση του θεμητού ανταγωνισμού, οπότε είπα πολύ ωραία, εντάξει, λογικό. Και μετά άρχισε να μιλάει και ο Επίτροπος και συνεχάρει βέβαια τους πάντες προτού καν ξεκινήσει η συζήτηση, περίεργο αυτό, και μετά άρχισε να μιλάει για κανόνες που θα ήθελε να θεσπίσει και άκουσα και όλη τη συζήτηση. Άρα αυτή τη στιγμή τι λέμε, ότι θα καταργήσουμε τις διμερείς συμφωνίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται και αναλαμβάνει αυτή την όλη διαπραγμάτευση και θα συνειδητοποιήσετε βέβαια ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες δίνουν επιδοτήσεις και ενισχύσεις στους αερομεταφορείς τους. Τι κάνουμε όμως εμείς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο μας απασχόλησε τελικά ήταν οι κρατικές ενισχύσεις. Επομένω, δεν ξέρω αν μιλάμε εδώ πραγματικά για ανταγωνισμό. Νομίζω ότι το πραγματικό μας θέμα ήταν οι κρατικές ενισχύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Έναν ακόμα ομιλητή έχουμε. Ο κύριος Κέρι θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως Ευρωβουλευτές φαντάζομαι ότι και εσείς θα επιβάζετε σε πτήσει πολύ περισσότερο από άλλου πολίτε και προφανώ μα ενδιαφέρουν οι αεροπορικέ μεταφορέ και προφανώ θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι σημαντικό για όλου, όχι μόνο για μα. Έτσι λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε δει πολλές εταιρείες low cost, όπως η Ryanair, με την οποία πετάω πολύ συχνά στο παρελθόν. Όταν δεν υπήρχε η Ryanair και ανάλογες εταιρείες, οι πτήσεις κόστιζαν πάρα πολύ ακριβά. Και έχουμε τώρα και άλλες εταιρείες, Erlingus και πολλές άλλες, οι οποίες ε, προτείνουν τιμές ε, ιδιαίτερα ανταγωνιστικέ. Ο ανταγωνισμό όμω θα πρέπει να ισχύει σε διεθνέ επίπεδο και έχουμε επιζήμιε αθέμητε πρακτικέ από τρίτε χώρε. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο ότι θα πρέπει όντω να ταχθούμε κατά των πρακτικών αυτών. Ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματο τώρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπο Έτιγκερ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Σημειώνω αυτά που είπατε και βλέπω ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία με το σχέδιο κανονισμού. Ο εισηγητής σας, ο κύριος Πίπερ, συμφωνείτε με αυτό το κείμενο που εκπονήθηκε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ορισμένοι συνάδελφοι ανέφεραν προβλήματα και βεβαίως έχουν δίκιο. Ο κανονισμός δεν πρόκειται να τα επιλύσει όλα τα προβλήματα αλλά είναι ουσιώδης πρόοδος στην πορεία προς έναν ισότιμο ανταγωνισμό προς το συμφέρον των αεροπορικών εταιριών που εδρεύουν στην Ένωση και επίσης προς το συμφέρον και όσων εταιριών τρίτων χωρών θέλουν να συμμετάσχουν ε, σε αυτόν τον ανταγωνισμό αλλά με ισότιμες συνθήκες και σε τελευταία ανάλυση προς το συμφέρον και των επιβατών άρα των καταναλωτών, των πολιτών που με αυτόν τον τρόπο θα πληρώσουν καλύτερες τιμές για υπηρεσίες καλού επίπεδου, θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ διαφόρων ανταγωνιστών και να κάνουν τις ε, πτήσεις τους. Είναι μια πορεία στην οποία ε, μια σαφής ε, ψήφος του Κοινοβουλίου θα συμβάλλει ιδιαίτερα. Και από πλευράς ε, της συναδέλφου Βούλτς ε, σας ευχαριστώ και τονίζω ότι το σχέδιο κανονισμού αυτού είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη μεγάλη κατεύθυνση για να έχουμε μια σωστή αγορά των αερομεταφορών. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε Λεοπρόεδρος. Και τώρα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Πίπα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αγαπητέ Αλφα είτε για την ενέργεια, είτε για τον ε, προπολογισμό, είτε τώρα για τι μεταφορές, είστε πάντα πιστικό. Ευχαριστώ του συναδέλφους που με ενεθάρναν με τι παρεμβάσει του και με στήριξαν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ευχαριστώ του και όλου των άλλων πολιτικών ομάδων, όλου του συνεργάτε των διαπραγματευτικών μα ομάδων, του βοηθού μα φυσικά. Όλου αυτού θέλω να τους ευχαριστήσω. Χαίρομαι που από ό,τι φαίνεται όλα τα κράτη-μέλη τη Ένωση ε, δρούν προ την ίδια κατεύθυνση και καταφέραμε λοιπόν να ε, κάποιες ε, ανησυχίες κάποιων μικρότερων χωρών που, ήθελαν, ε, που φοβόνταν ότι δεν θα υπήρχαν ε, ε, εάν υπήρχαν συγκρούσεις θα υπήρχε κίνδυνος να μην υπάρχουν επαρκείς πτήσεις. Ο κανονισμός αυτός θα ήταν πιο ισχυρός εάν μπορεί να παρέμβει εάν υπάρχει κίνδυνος να υπάρξουν αθέμητες πρακτικές. Ε, αυτή είναι η διαφορά με τον παλιό κανονισμό 868, ο οποίο στην ουσία δεν ε, εφαρμόστηκε αύριο. Λοιπόν, νομίζω θα είναι μια καλή μέρα για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε, μια καλή μέρα για μια Ευρώπη που μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της. Αν δρούμε από κοινού στην Ευρώπη, στην Ένωση, μπορούμε να υπερβούμε του εγωισμούς κάποιων ε, επιχειρηματικών τομήλων και κάποιων εθνών. Οπότε σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ο πρόεδρο, κύριε Πίπερ. Κλείνει η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έκθεση Χολμάιερ όσον αφορά τις κατευθύνες γραμμές για τον προπολογισμό του 2020, τμήμα 3. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια, λοιπόν, την κυρία Χολμάιερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, ευχαριστώ επίσης πολύ τους σκιώδεις συναδέλφους οι οποίοι ασχολήθηκαν τόσο πολύ, έκαναν τόση πολύ δουλειά, ούτως ώστε να έχουμε σωστές κατευθύντηρες γραμμές, να καθορίσουμε τις προτεραιότητές μας για το 2020, δεν ήταν ε, απλή προσπάθεια γιατί δεν είναι απλή η χρονιά αυτή. Θα είναι η τελευταία χρονιά των τελευταίων ε, προοπτικών και πρέπει να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση προς, το, προς τη νέα περίοδο. Και δεν είναι απλή χρονιά γιατί έχουμε και το θέμα του Brexit. Οι οποίες πάνε από το μια καταστροφή στην άλλη οι για τον Brexit και δεν έχουμε ιδέα τι θα προκύψει. Και επίσης, διότι έχουμε ενώπιον μας μεγάλες ε, προκλήσεις, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, κοινωνικές συνθήκες, ευημερία. Έχουμε προκλήσεις επίσης ε, για την αναπτυξιακή μας βοήθεια και για τα θέματα των μεταναστευτικών ροών, των ανθρώπων δηλαδή που ζουν ε, πολύ χειρότερα από εμά σε τρίτες χώρες και έχουμε το θέμα της ασφάλειας εσωτερικής και εξωτερικής. Θέλουμε δηλαδή με τον καλύτερο τρόπο να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Αγαπητέ συνάδελφε, έχω ένα αγαπητέ συνάδελφε κύριε Επίτροπε, στον τομέα του έρασμος και της νεότητας σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ να δεχτείτε τα αιτήματά μας γιατί πιστεύω ότι μόνο αν οι νέοι και γενικότερα εργαζόμενοι έχουν καλές θέσεις εργασίας αν έχουμε μια οικονομία που να μπορεί να προσφέρει καλές θέσεις εργασίας και αν μπορέσουμε να επενδύσουμε στις τεχνολογίες του μέλλοντος πρέπει να καταρτήσουμε τους νέους μας. Και θέλουμε, στα πλαίσια της κατάρτισής τους, να μπορούν να επισκεφτούν και άλλες χώρες, να γνωρίσουν άλλες χώρες, ε, τις γειτονικές τους, να έχουν στενές επαφές. Τα προγράμματα λοιπόν αυτά πρέπει να ενισχυθούν. Υπάρχουν προγράμματα όπως το Horizon Ευρώπη, όπου είναι χαμηλό το ποσοστό επιτυχίας ε, ε, τα λέω αυτά επανειλημμένα, ίσως σας κουράζω. Κι εγώ όμως κουράζομαι που τα λέω. Προγράμματα όπως το COSME, όπως το πρόγραμμα για τις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπου έχουμε απορρίψεις 97%. Όχι γιατί είναι άσχημα τα προγράμματα που υποβάλλονται, γιατί δεν υπάρχουν ε, επαρκή πόροι. Δεν έχουν δεχθεί τα κράτη-μέλη επαρκή πρικοδότηση των προγραμμάτων αυτών. Πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους να αποκτήσουν θέσεις εργασίας που να έχουν μέλλον όπου να αισθάνονται ασφαλείς. Να είναι θέσεις εργασίας που θα διατηρηθούν και στο μέλλον και οι εταιρείε που τις προσφέρουν να μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις για να συνεχίσουν να εργάζονται. Αυτό είναι το βασικό καθήκον. Αυτά είναι τα καθήκοντα που πρέπει να ε, επιτελέσουμε. Να έχουμε νέους εργαζόμενους ε, σωστά καταρτισμένους και οι θέσεις εργασίας να μπορούν να στηριχθούν και να στηρίξουμε και την καινοτομία να είναι θέσει εργασία δηλαδή που θα έχουν και μέλλον, που θα μα διατηρήσουν ανταγωνιστικού. Να μπορέσουμε να αντέξουμε τον ανταγωνισμό των άλλων τμήματων του κόσμου. Και να το πω απόλυτα ανοιχτά, ελπίζω τα κράτη-μέλη να μην έχουν ε, την στάση που έχουν τις τελευταίες μέρες. Ε. Το Συμβούλιο δεν είναι βέβαια παρόν, αλλά πρέπει να το τονίσω. Δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε τελευταία στιγμή με στη νύχτα πρέπει από νωρί να συμφωνήσουμε επί του περιεχομένου ακόμη και αν όλα τα θέματα αυτά θα ε, αποφασιστούν στην επόμενη ε, θητεία μας πρέπει να συζητήσουμε με το Συμβούλιο να μας πει την άποψή του και θα ήθελα και η Επιτροπή να μας θέσει τις προτεραιότητές της. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφε. Το λόγο τώρα εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ο Επίτροπος Έτιγκερ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με τη συζήτηση σήμερα ξεκινάτε τις συζητήσεις για τον προπολογισμό για το έτος 2020 που θα είναι μια ε, ιδιαίτερη χρονιά. Πρώτα απ' όλα είναι η τελευταία χρονιά της ε, πολιτούς περίοδου 14-20 από την άλλη πλευρά. Υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα για τον Brexit Κανείς δεν ξέρει. Εάν οι συνάδελφοι από το Ηνωμένο Βασίλειο και η χώρα δηλαδή θα συμμετάσχει πλήρως στο δημοσιονομικό πλαίσιο εάν θα εφαρμόσουν δηλαδή αυτά που αποφασίστηκαν το 2013 ομοφόνο στο Συμβούλιο και το τρίτο θα έχετε νέα θητεία εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και νέα επιτροπή. Πρέπει λοιπόν ε, να συμβάλλουμε όσο μπορούμε για όλους αυτούς τους λόγους στο να υπάρξει σταθερότητα, τόσο ώστε τα προγράμματα για την ανάπτυξη Ευρώπης να μπορέσουν να συνεχίσουν να δρουν θετικά και οι κοινοί μας στόχοι να λάβουν την αναγκαία χρηματοδότηση και να επιτευχθούν. Ευχαριστώ την κυρία Χολμάια για την ε, θαυμάσια προεργασία της, η οποία προσπαθεί να συνδυάσει τις διαφορετικές ε, προσδοκίες των συναδέλφων και των πολιτικών ομάδων, να τα φέρει όλα αυτά σε ένα κοινό παρονομαστή. Αυτό καμιά χρονιά δεν είναι εύκολο και σε μια εκλογική χρονιά είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους οι οποίοι ήταν διατεθειμένοι να, συνεργάσουν, να συνεργαστούν όχι να κάνουν ε, προεκλογικές διακηρύξεις, να συνεργαστούν ουσιοδός. Ευχαριστώ, γιατί οι στόχοι του Κοινοβουλίου βασικά είναι και οι στόχοι της Επιτροπής. Έχουμε αυτή την αλλαγή. Νέο Κοινοβούλιο. Είστε αρμόδιοι για τη θέση του Κοινοβουλίου και ελπίζω και το επόμενο Κοινοβούλιο να μην έχει αντιδιαμετρικά διαφορετική άποψη, να βασιστεί στη δική σας θέση. Ελπίζω πολύ στο Κοινοβούλιο να παραμείνουν, ιδιαίτερα αυτοί που είναι αρμόδιοι για τη δημοσιονομική πολιτική. Δηλαδή να επανεκλεγούν. Από την εισηγήτρια μέχρι πολλούς άλλους οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα προπολογισμών, με τις ικανότητές τους. Και ελπίζω να μπορέσουν να συνεχίσουν να βοηθούν και στην επόμενη θητεία. Βέβαια και τι θα γίνει με την Επιτροπή και αυτό πολύ συναρπαστικό θέμα. Γιατί η περίοδος συνδιαλλαγής θα ξεκινήσει στις 19 Οκτωβρίου. Δηλαδή με την παρούσα Επιτροπή. Και τελειώνει στις 18 Νοεμβρίου. Ίσως ε, με την επόμενη Επιτροπή. Είτε ίσως αν χρειαστεί να παραμείνει περαιτέρω η παρούσα Επιτροπή γιατί δεν θα γίνει αποδεκτή εγκαίρως ε, η επόμενη, τότε το βασικό είναι να υπάρξει ε, συνέχεια στη δουλειά μας για να διασφαλίσουμε την ε, σταθερότητα στην Ευρώπη που έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια γέφυρα προς την ε, μελλοντική Ευρώπη, να επενδύσουμε στους πολίτες την καινοτομία και την ασφάλεια. Αυτός είναι ο τίτλος τον οποίο επέλεξε η κυρία Χολμάιερ. Ιδιαίτερα κατάλληλος, θεωρώ, γιατί οι πολίτες πρέπει να πιστούν για την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης και να υπάρχει γι' αυτό επαρκής χρηματοδότηση. Όπως και πριν, οι κοινέ μας προτεραιότητες είναι η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και καλύτερες ηθίκες ζωής, έρευνα, η νέα γενιά, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να συμβάλλουμε στο να υπάρξει περισσότερη ανταγωνιστικότητα και οικονομική ανάπτυξη. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Τα τελευταία έξι χρόνια σε γενικές γραμμές ήταν καλά χρόνια για την ευρωπαϊκή οικονομία. Χρόνο και χρόνο αυξανόταν, ε, αυξάνονταν ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης και ήταν υψηλότερος από ό,τι είχε προβλεφθεί. Υπήρξαν περισσότερα φορολογικά έσοδα από όσα προβλέπονταν. Κάθε χρόνο μειωνόταν η ανεργία. Αυξάνονταν θέσει εργασία και μειωνόταν και η ε, ανεργία των νέων. Βέβαια, κατά πολύ απέχουμε ακόμη από μια ικανοποιητική κατάσταση. Τα τελευταία 6 χρόνια ήταν καλά χρόνια και με βάση όλε τι ε, προγνώσει ε, αρχίζει να μειώνεται αυτή η θετική εξέλιξη. Γι' αυτό ο προπολογισμό 2020 πρέπει να μας δώσει τα κατάλληλα εργαλεία κατά της ύφεση, κατά της στασιμότητας, κατά των κρίσεων ούτω ώστε να υπάρξει περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερε θέσει εργασία, περισσότερη ευημερία, ανταγωνιστικότητα στα πλαίσια των περιορισμένων ε, ε, πόρων που διαθέτουμε για το κόσμο και τις μικρομεσαίες μας για να ε, προωθήσουμε καινοτόμες αντιλήψεις για το έρασμο συν για να αυξήσουμε τις διαπολιτιστικέ μας δυνατότητες, για την κυβερνοασφάλεια, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της φύσης. Έχουμε μια σειρά από προγράμματα που πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση και που με βάση τους περιορισμένους πόρους μας πρέπει να τα ενισχύσουμε. Γι' αυτά χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη ευελιξία. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει από κοινού εν μέρη κατά του Συμβουλίου να παλέψουμε για να υπάρξει περισσότερη έγκαιρη ευελιξία για να μπορούμε να αντιδράσουμε στις προκλήσεις που θα έχουμε εντόπιόν μας, ενώπιόν μας και στα καθήκοντα που θα έχουμε. Πρέπει να προσέξουμε, ιδιαίτερα στην πολιτική συνοχής, να υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις πληρωμών όλα όσα είχαμε ως υποχρεώσεις να καλυφθούν τώρα ως πληρωμές. Για να μην έχουμε τα επόμενα χρόνια ε, ε, μεγάλες μεταφορές πιστώσεων. Το Συμβούλιο στο ΕΚΟΦΗΝ αποφάσισε τις καθεντήριες γραμμές στις 12 Ιανουαρίου. Σήμερα και τις επόμενες μέρες θα υποβάλλετε εσείς τις προτεραιότητες και τις καθεντήριες γραμμές σας ως ε, δεύτερο σκέλος της ε, ε, αρμόδιας αρχής για τον προπολογισμό, εμείς ως Επιτροπή θα κάνουμε τις αναγκαίες ενέργειες για να συνδυάσουμε τις εργασίες των δύο αυτών. Ο πρώτος τριμερής διάλογος θα είναι στις 20 Μαρτίου, θα είναι η πρώτη ευκαιρία. Επαναλαμβάνω, οι προτεραιότητές σας είναι σχεδόν ταυτόσιμες με τις δικές μας. Σας ευχαριστώ για την καλή αυτή προεργασία. Σας ευχαριστώ που όλοι επιδείξατε ότι δεν ήσασταν διτεθειμένοι να μπερδέψετε την προεκλογική στρατεία με την αναγκαία προεργασία σας για τον προπολογισμό του 2020 για να κάνετε ό,τι μπορείτε για τους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τις παρεμβάσεις εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Το λόγο εξ ονόματος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λεκού Κόμματος έχει ο κύριος Κέλλη για τρία λεπτά. Κύριε Κέλλη, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια στην κυρία Χολμάιρ. Καθώς επίσης και τον Επίτροπο κύριο Ότι που κάνει τόσο πολύ καλή δουλειά σε αυτό το χαρτοφυλάκιο όπως και στο προηγούμενο. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι, το, είναι σημαντικό ο προπολογισμό του 2020 να θέσει τη σωστή κατεύθυνση για το επόμενο πολιτεία δημοσιονομικό πλαίσιο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιε είναι οι βασικέ προτεραιότητε για την επόμενη δεκαετία. Θα πρέπει να έχουμε ισχυρό προπολογισμό, καλά χρηματοδοτημένο και να ε, είναι ένα προπολογισμό που θα κοιτάει το μέλλον, όπω είπε ο Επίτροπο. Χαίρομαι που εστιαζόμαστε στην έρευνα και την καινοτομία. Το έχουμε επανειλημμένο στο μίση, το μίση είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να συνεχίσει να αναπτύσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δημιουργούνται θέσει εργασία σε 27 χώρε και να βελτιωθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μα. Καλωσορίζουμε την έμφαση που δίνει ο εισηγητή σε προγράμματα όπω Horizon 2020, το κόσμο και οι ψηφιακέ επενδύσει. Δεύτερον, καλωσορίζω τη σημασία που δίνεται στην κλιματική πρόκληση. Είναι σημαντική πρόκληση στο μέλλον για να διασφαλίσουμε ε, ότι θα εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει στην αιχμή του δωράτου της κλιματικής δράσης. Ήδη, κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής της Κομισιόν, ε, έδειξε σημαντική, ε, σημαντικό ηγετικό ρόλο με κορονίδα το Παρίσι του 2015. Αυτά τα προγράμματα είναι πολύ σημαντικά και νομίζω ότι θα μπορέσουμε σε αυτό να χρηματοδοτήσουμε τις απαραίτητες δράσεις. Είναι, πολύ πετυχημένοι τα τελευταία χρόνια. 35.750 γιγα, ώρες, ε, ήταν η παραγωγή τη ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων το 1% ε, ήταν... Ε, ε, απονεώνωση ενέργεια στην Ιρλανδία. Το πρόγραμμα Invest EU, επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επίση ήταν πολύ σημαντικό και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τριμερή διάλογο. Χρειαζόμαστε ένα καλά χρηματοδοτημένο προπολογισμό και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε το 2020 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συζητήσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Τέλος, συμφωνώ με τον Επίτροπο που αναφέρθηκε στο Brexit. με αποτέλεσμα 308 ψήφους υπέρ, 302 κατά, αποφασίστηκε στο κοινοβούλιο μας ε, να μην ε, βγούμε ε, ατακτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χαίρομαι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει έτοιμα μπλε κάρτα από την κυρία Νιριάντα. Τη δέχεστε? Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε το λόγο. Καλώ ορίζω το γεγονό ότι δείχνει τόσο πολύ σημασία σε κλιματικά ζητήματα. Όμως ένα πολύ μικρό ποσοστό του προπολογισμού αφιερώνεται στο κλίμα. Το ερώτημα είναι γιατί η δική σου ομάδα αρνήθηκε να μιλήσουν άνθρωποι για το εγκληματική αλλαγή στον Πρωθυπουργό σας. Γιατί συνεχώς ε, ψηφίζετε υπέρ υπέρ της χρηματοδότησης των ορυκτών υδρογονανθράκων αντί ε, να μετακινηθούμε προς ε, πιο φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Μπορείς να μας το εξηγήσεις αυτό. Ε, ε, ε, μπορώ να απαντήσω παρόλο που είναι πολιτική πρόκληση αυτό που λέτε. η ομάδα μου ε, και εγώ ίδιος έχω εκπροσωπήσει το Κοινοβούλιο ε, στο συζητήσεις του Παρισιού ε, οπότε και έχω, ήμουν και εισηγητή σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον οπότε οι περγαμηνές μου είναι σαφείς δεύτερον το, το κόμμα μου είναι κυβερνά αυτή τη στιγμή και έχουμε ένα καινούριο υπουργό που αυτή τη στιγμή προετοιμάζει το σχέδιο ενέργειας και κλίματος, το οποίο θα είναι πάρα πολύ φιλόδοξο. Το, το ίδιο και οι στόχοι του, για το 2040, 25% για την κλιματική δράση. Οπότε και το Fiona Γκέιλ, το κόμμα μου, και η κυβέρνησή μας, αλλά και το ΕΛΚ εδώ πέρα, ηγούνται τις προσπάθειες, προσπάθειες προκειμένου ε, να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή με πρακτικό τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εξ ονόματο τη Προδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το λόγο έχει η κυρία Ντουανέκ Μογά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με μεγάλη χαρά Μιλώ εξ ονόματο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για τον προπολογισμό του 2020, την εκπόνηση του προπολογισμού αυτού που είναι ο τελευταίο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου που πάει μέχρι το 2020.